τις ανησυχίες του κυρίου Φερέρα, τις ανησυχίες που τονίσατε μετά από όλες τις καταστροφές που γνωρίσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα για την εισήγησή σας. Θα έχουμε την ψηφοφορία αύριο στις 12. Τώρα έχουμε την τελευταία έκθεση, την και έκθεση της κυρίας Θεοχάρους σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ο δρόμος της προόδου. Έχετε τέσσερα λεπτά κυρία εισηγήτρια. Πρόεδρε, είναι παραδεχτό πως η Αφρική κυρίως αλλά και πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη που μαστίζονται τόσο από τη φτώχεια όσο και από τα δημοκρατικά ελλείμματα αποτελούν το μαλακό υπογάστριο του διεθνού συστήματος. ανέλαβα να εκπονήσω με τη συνδρομή βεβαίω ε, όλων των πολιτικών ομάδων την έκθεση αυτή πιστεύοντας ακράδαντα ότι η ευρωπαϊκή ένωση μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της φτώχειας με πολλούς τρόπους και κυρίως με τη δημιουργία θέσεων εργασία και βεβαίω η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να βοηθήσει τον μισό περίπου πληθυσμό του πλανήτη που ζει κάτω από το όριο τη φτώχεια, έχοντα υπόψη την έλλειψη εμπιστοσύνη και την καχυποψία των λαών των υποαναπτύκτων χωρών προ τι αναπτυγμένε, αλλά και την πιθανή αντίδραση των λαών τη Ευρώπη για τη συνεχή αιμορραγία τη χρηματοδότηση των φτωχών προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε ευθύ εξ αρχή ότι η ανάπτυξη του τρίτου κόσμου θα αποτελέσει σημαντική ωφέλεια για την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση τρόπο βεβαίω. για παράδειγμα με την ανάπτυξη θέσεων εργασία μπορεί να αντιμετωπιστεί η μη ελεγχόμενη μετανάστευση και παράλληλα θα μειωθεί η αστάθεια στι φτωχέ χώρε. Βεβαίω, έχοντα υπόψη επίση ότι η βασική προπόθεση για την ανάπτυξη είναι η εγκατάσταση η αποκατάσταση και η βελτίωση τη δημοκρατία και των δημοκρατικών θεσμών και η λειτουργία ινστιτούτων εκδημοκρατισμού και φυσικά η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών καθώς επίσης και η δράση και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών καταγράψαμε ως ιδιαιτέρως σημαντικό και τον παράγοντα αυτό. δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην βελτίωση της εκπαίδευσης και στην ελεύθερη επιλογή για παραμονή των επιστημόνων και των εξειδικευμένων επαγγελματιών στις χώρες τους. η πανδημία του aids και οι συμπαρομαρτούσες καταστάσεις ως ιδιαιτέρως επιβαρυντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διαιώνιση του φαύλου κύκλου της φτώχειας ελήφθησαν ιδιαίτερω υπόψη και κατεγράφησαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι παραγόντε, ώστε να μην συνιστούν τροχοπέδι στην ανάπτυξη και στην ε, αντιμετώπιση της φτώχεια. Τέλος, λάβαμε υπόψη τις πολλαπλές προσπάθειες που κατεβλήθησαν ανεπιτυχώς από την παγκόσμια κοινότητα, αλλά και όλε τι διεθνείς συμβάσει με τι οποίε προσπάθησε ο κόσμο να αντιμετωπίσει τη φτώχεια κατετέθησαν 97 τροπολογίες και καταφέραμε να φτάσουμε σε συνενετικές προτάσεις σε πολλές από αυτές. Παραμένουν κάποιες ιδεολογικού μάλλον χαρακτήρα τροπολογίε τροπολογίες τις οποίες δεν έχουμε, πλήρη, ε, συμφωνήσει, δεν έχουμε πλήρως για όλα και κάποια τυπικά ζητήματα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία γιατί αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το ΚΑΤΣΔΙ. Έχουμε αρκετούς ομιλητές. Η πρώτη κυρία Μπασέσκου, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, με την τωρινή οικονομική κρίση η οποία οδηγεί σε μία αύξηση των τιμών τροφίμων και καυσίμων υπάρχουν πολλά άτομα που οδηγούνται στη φτώχεια. Είναι μεγάλη πρόκληση για τις υποανάπτυξη χώρες ακόμη και αν στην ε, Ευρώπη η οποία είναι μεγάλη δύναμη ε, ε, δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος και θα πρέπει να βρούμε καινοτόμες μεθόδους χρηματοδοτήσεως του τρίτου κόσμου και να καταπολεμήσουμε στην φτώχεια σε αυτές τις χώρες. Ελπίζω ότι ε, στη διάσκεψη κορυφής για την επίτευξη των στόχων της χιλιετηρίδας που οργανώνεται τώρα θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε νέες μεθόδους επιλύσεως του αγώνα κατά της φτώχειας. Γι' αυτό και η χώρα μου ε, έδωσε μία βοήθεια 100 εκατομμυρίων ευρώ στην ε, Μολδαβία υπομορφή δωρεάς. Θα ήθελα να σας πω ότι ουσιαστικά στην διαδικασία αυτή, ε, στο Catch the Eye δηλαδή, θα έχουμε ακόμη τέσσερις ομιλητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ιδίω ευχαριστώ για την γενεοδορία τον Πρόεδρο, αλλά θα είμαι σύντομος. Αναφέρομαι στην Γεωργία, γιατί η Γεωργία όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και την προμήθεια τροφίμων έχει βασικό ρόλο. Χρειάζεται μία σταθερή γεωργία, αλλά χρειάζεται και μία σταθερή τιμή των προϊόντων στη διεθνή αγορά για να μπορέσει να υπάρχει μία λειτουργική ε, γεωργία στις υποανάπτυξη χώρες και χρειάζονται και ε, σταθερές πολιτικές συνθήκες και καταπολέμηση της διαφθοράς για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να μειωθούν η φτώχεια. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, ε, είδαμε ότι οι επιδοτήσεις, οι εξαγωγικές ευρωβογές της ευρωπαϊκής πολιτικής απεδείχθησαν εσφαλμένες και θα πρέπει να καταργηθούν. Ο κύριος Νικολάσιτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Οι επενδύσεις είναι επενδύσεις ε, για την γενικότερη ανάπτυξη των χωρών ε, εάν επενδύουμε στους ε, δημόσιους οργανισμούς και στα άλλα θεσμικά όργανα κάθε φτωχής χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς δεν σέβεται το γεγονός αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν γέννη και δεν δίνουν ε, το ελάχιστο της εκατό το οποίο προβλέπεται για την ε, υγεία. Εγώ θεωρώ ότι η υγεία και η παιδεία, κυρίως ε, η βασική εκπαίδευση, θα πρέπει να αποτελούν τη βάση οποιασδήποτε μορφής πολιτικής. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις δαπάνες προς αυτούς τους δύο τομείς. Θα πρέπει να επενδύουμε περισσότερο. Ε, στους δύο αυτούς τομείς, στην υγεία και στην ε, ε, παιδεία, γιατί αυτή είναι η πιο βασική. Και τέλος ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μείωση της ένδυας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε χώρες στη φάση ανάπτυξης σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μία στοχευμένη πολιτική για την ανάπτυξη και θα πρέπει να βοηθήσει την αυτόνομη ανάπτυξη και την κυρίαρχη ανάπτυξη των χωρών αυτών. Ε, η προσπάθεια να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διορθώσεις στις ελλείψεις που υπάρχουν επί του θέματος αυτού. Το σύστημα υγείας, ε, ένα υγειονομικό σύστημα καλού επίπεδου, η ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, η διατροφική ανεξαρτησία και ασφάλεια, μόνο αυτά θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη μείωση της ένδυας. Αν δεν υπάρχουν σωστές και ισότιμες εμπορικές σχέσεις, πέραν οποιοδήποτε κανόνα δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις αποσχόλησης οι οποίες θα είναι διαρκείας. Λυπάμαι ε, διότι συνεχώς αγνοούμε ε, ότι επιβάλλονται δεσμεύσεις ε, στις χώρες, στις αναπτυσσόμενες χώρες και δεν ξεχνάμε το χρέος. Η μείωση του χρέους είναι πάρα πολύ σημαντική για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ευχαριστώ και τώρα ο λόγος στον Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντοτε εξ ονόματος της συναδέλφους κυρίας Γιώργεβα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Θεοχάρους για αυτήν την πλήρη έκθεση ισορροπημένη. Πάνω σε ένα θέμα επικαιρότητα είναι ένα από τα θέματα το οποίο ε, συζητείται στο υψηλότερο επίπεδο των διεθνών ηγετών στα Ηνωμένα Έθνη. Τονίζεται δικαίως ε, μια ε, μεγάλη ανησυχία που διατρέχει την διεθνή συνεργασία, την μείωση της πτώχειας, την δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι κάτι το κατεπήγον λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των τιμών πετρελαίου και πρώτων ύλων, όπως είπατε κυρία Μπαζέσκου, ορισμένα τρόφιμα και αυτό με ανησυχεί στις χρηματοπιστωτικές ε, ε, υπηρεσίες ότι υπάρχει κερδοσκοπία, υπερκερδοσκοπία στις πρώτες σύλλες με τον κύριο Τσόλο σήμερα το πρωί ε, συζητήσαμε στις Βρυξέλλες και δεσμευθήκανε πέραν των όσων παρουσίασε αυτή την εβδομάδα για την ρύθμιση των παραγόγων να θεσπίσω μέσα για τον έλεγχο και την μείωση της κερδοσκοπίας που είναι σκανδαλώδης ε, στις πρώτες ύλες, κυρίως τις αγροτικές, εις βάρος των χωρών που έχουν λιγότερη αυτονομία όσο προς την επισητιστική επάρκεια. Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η κοινωνική πολιτική είναι σημαντικά θέματα για την μείωση της ένδυας, για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντικτύπου ε, του κοινωνικού. Υιοθετήσαμε τον Απρίλιο μια ανακοίνωση με δέσμευση να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να υπερνικήσουν την κρίση. Το Συμβούλιο στήριξε αυτήν ε, την ε, πρωτοβουλία, αυτό δείχνει τη δέσμευση για την απασχόληση και μια πρόοδο κοινωνικής ε, προστασίας για τους πιο ευάλωτους. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο αμυντικοί στις κρίσεις, αλλά να δρούμε μακροπρόθεσμα. Νομίζω, κύριε Φερέρα, ότι αυτό ήταν και το νόημα της παρέμβασής σας. Να δράσουμε για τους πιο αδύναμους μακροπρόθεσμα. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δεσμευσή τους για τις, τους τη για την ανάπτυξη και υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη μια σύνοδο για το θέμα αυτό, η προώθηση της απασχόλησης των πολιτικών κοινωνικής προστασίας που ο κύριος Νικολαϊσέσκου ανέφερε περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε ένα σημαντικός πυλώνας των ε, στόχων της χιλιετίας η Κομισιό είναι πεπισμένη ότι δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί η ένδια χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις δύο αυτές απόψεις και όπως τονίσατε πολύ καλά κυρία εισηγήτρια θα πρέπει οι πιο ευάλωτοι να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας των αναπτυξιακών. Βεβαίως οι πολιτικές μας δεν έχουν αξία αν δεν υλοποιούνται, αν μείνουν στα λόγια χρειάζεται μια θέσπιση ε, ad hoc ε, για ευελιξία με τον τρόπο με τον οποίο οι δωρητές ε, μπορούν να στηρίξουν το επίπεδο των δαπανών στον κοινωνικό τομέα και την επισητιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει τους πιο αδύναμους στην ικανότητα παραγωγής γεωργικής για να μπορέσουμε και να στηρίξουμε την κυριαρχία, την αυτονομία, δεν θα έλεγα την αυτάρκεια, την αυτονομία των χωρών αυτών σε περιφερειακό επίπεδο. Ο συνάδελφος Κιμπάλστα στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής υποστηρίζει τις προσπάθειες αυτές. Η έκθεσή σας τονίζει δικαίως, κυρία εισηγήτρια, τη σημασία της ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών ε, για μια πρεπή εργασία του ε, Παγκόσμιου Συμφώνου για την Απασχόληση. Υποστηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και συμφωνώ πλήρως μαζί σας κυρία Θεοχάρους για να πω ότι θα πρέπει να εκπονήσουμε μια θεώρηση ευρωπαϊκή για την κοινωνική προστασία. Έχουμε αρχίσει προκαταρκτικές εργασίες που θα οδηγήσουν σε αυτήν την, το κοινό όραμα, την κοινή θεώρηση. Ε, θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Ανάπτυξη 2010 που θα αναφέρεται στην κοινωνική προστασία και πρόνοια στις ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει να βρούμε καινοτόμες λύσεις. Νομίζω ότι οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να προσφέρουν εν μέρη αυτές τις καινοτόμες λύσεις. Σας ευχαριστώ που επισύρετε την προσοχή μας πάνω στο σημαντικό ρόλο της ισότητας των φύλων για τη μείωση της φτώχειας. Τα κρατημέλη ακολουθούν αυτή τη γραμμή και για το λόγο αυτό στις 14 4 Ιουνίου το Συμβούλιο θέτησε ένα πρόγραμμα δράσης για να υποστηρίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ισότητα μεταξύ των φύλων και την προσάρτησε ε, στα συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα όσον αφορά στους στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ την κυρία Θεοχάρους. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Ε, λύεται η συνεδρίαση.